Και αν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση στα πρακτικά, θα θεωρήσουμε ότι έχουν επιβεβαιωθεί αυτοί οι διορισμοί. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος μας έχει δώσει ένα διορθωτικό σε ένα κείμενο του Κοινοβουλίου, το ίδιο και η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Και σύμφωνα με το άρθρο 216 γίνουν αποδεκτά ε, όταν γίνεται ένα αίτημα από μια πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον 40 μέλη. Ε, στην ιστοσελίδα ε, η Ολομέλη Απευθείας θα δείτε το σχετικό τίτλο που έχουμε δημοσιεύσει για τα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης. Το Κοινοβούλιο τον Ιούλιο μαζί